Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής ΕΚΟΝ για το 2019. Με ιδιαίτερη χαρά θα προεδρεύσω σήμερα το πρωί, αλλά είμαι ταυτόχρονα και συγκήτρια στην πρώτη έκθεση και Ω συντονίστρια θα διαβάσω και τα σχόλια πολλών σχεδόν εισηγητών σήμερα το πρωί, οπότε θα σας κουράσω, θα μου ακούτε συνέχεια και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη. Αλλά αυτά έχει η ζωή. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω καλωσορίζοντάς σας και να σας προτείνω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη όπως έχει κυκλοφορήσει στο δεικτικό χρονοδιάγραμμα. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν παρατηρήσεις, θα ήθελα παρακαλώ να εγκρίνουμε αυτό το δεικτικό χρονοδιάγραμμα και τη σχετική ημερήσια διάταξη. Περνάω τώρα στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης την έγκριση των πρακτικών δηλαδή. Στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα θα δείτε ένα μακροσκελή κατάλογο με πρακτικά συνεδριάσεων. Δεν πρόκειται να διαβάσω όλο τον κατάλογο. Θα ήθελα παρακαλώ να τα εγκρίνουμε όμως αυτά τα πρακτικά. Δεν βλέπω αντιρρήσεις, οπότε εγκρίνονται όλα τα πρακτικά. Και περνάμε στο σημείο 3 της ανακοινώσης του Προέδρου ή της Προέδρου, προκειμένου. Δύο ανακοινώσεις έχω εδώ. Στις 14 Ιανουαρίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, ε, η προγραμματισμένη συνεδρίασή μας για το απόγευμα της Δευτέρας και που περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα του 2019, ακυρώνεται. Δεν θα συνεδριάσουμε δηλαδή στο Στρασβούργο ή ΕΚΟΝ τη Δευτέρα. Επίσης, 3η ε, 22 Ιανουαρίου θα έχουμε οικονομικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Νάντια Καλβίνο, την Ισπανίδα Υπουργό Οικονομίας και Επιχειρήσεων, επαναλαμβάνω 22 Ιανουαρίου, 2.30 με 4 το απόγευμα. Αυτά τα δύο σημεία έχω σαν ανακοινώσει. Το επόμενο σημείο, το σημείο 4 της ημερήσης διάταξης, είναι η ενημέρωση για τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις και έχω αρκετές πληροφορίες εδώ. Καταρχήν, δια, τριμερής διάλογος 13, 13 Δεκεμβρίου, ΠΕΠ, τρίτη, τρίτος για τα ΠΕΠ έγινε και συμφωνήσαμε καταρχήν πολιτικά για τα εκκρεμή θέματα όπως την έγκριση ΠΕΠ από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ε, της παρεμβάσεις της ΕΙΟΠΑ, κάποιες επιλογές ε, διαχωρισμού και η οριστικοποίηση του σχεδίου συμφωνίας ε, συνεχίζεται. Θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Δεύτερη ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο για το μηχανισμό προστασίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στις 18 ε, Δεκεμβρίου ήδη ελήφθη πολιτική συμφωνία στον πρώτο τριμερή διάλογο για τον πιθανό μηχανισμό προστασίας με ο χρονοδιάγραμμα που ισχύει άσχετα με το πώς ε, πυροδοτούνται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μάλιστα για τα τυλοποιημένα έχουμε τρία χρόνια και για τα μη τυλοποιημένα ανάλογα με τις εγγυήσεις ε, πολύ περισσότερα, 29. Πάντως, ε, ε, ένα χρόνο θα υιοθετηθεί ένα συνολικό μηχανισμό προστασία. Και στι 7 Ιανουαρίου, η Κορεπέρ συμφώνησε σε ένα κείμενο και η ε, επαναδιαβούλευση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ θα γίνει 21 και 22 Ιανουαρίου τρέχοντο έτου. Και τέλο, την τριμερή διάλογο τη 8 Ιανουαρίου για τα funds πρώτη, πρώτος τριμερής διάλογος για, τα, για τη διασυνοριακή κατανομή των συλλογικών αυτών αμοιβαίων κεφαλαίων και ο επόμενη, ε, επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει 5 Φεβρουαρίου. Ε, για τις ε, κοινοποιήσεις, για, τις, ε, για το pre-marketing των AIF, για τα ΟΣΕΚΑ, για τα τέλη, αξιολόγηση και αναθεώρηση και το τεχνικό, οι δήμονες έχουν λάβει την εντολή να συνεχίσουν τη διαπραγματεύση για τα αναπομείναντα ε, θέματα. Τώρα, περνάμε στη δική μου γνωμοδότηση την εισαγωγή τη πληροφορική τη διακίνηση και του ελέγχου των αγαθών που υπόκειται σε ειδικού ε, φόρου κατανάλωση. Ω εισηγήτρια, λοιπόν, θα ήθελα να σα ενημερώσω για λίγα λεπτά για το συγκεκριμένο θέμα. Μέχρι στιγμής ε, δεν ε, βλέπω όλους και ηγητές των πολιτικών ομάδων, γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τις πολιτικές ομάδες να ορίσουν τους και ηγετές τους για το θέμα αυτό. Είναι η πρόταση αυτή ένα τμήμα του πακέτου τεσσάρων προτάσεων του 2018 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα πακέτο νέων κανόνων για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης με τις γενικές ρυθμίσεις και τις ειδικού φόρους κατανάλωσης για τα εναπνευματόδη και τις ρυθμίσεις για την ε, εισαγωγή τη πληροφορική στη διακίνηση και του ελέγχου των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικού φόρου κατανάλωση. Συμφωνώ με το περιεχόμενο τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω εκ τούτου σα προτείνω να την εγκρίνουμε χωρί τροποποιήσει. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα και δεν θεωρώ ότι έχει δεν είναι επίμαχο πολιτικά και δεδομένου του φόρτου εργασία τη Επιτροπή και του ελάχιστου χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μα, θα σα πρότεινα, αν φυσικά δεν έχετε αντίρρηση και εσεί και οι σχεδόν να προχωρήσουμε με την απλοποιημένη διαδικασία με βάση τον εσωτερικό μας κανονισμό. Και αν συμφωνείτε θα παρουσιάσω την έκθεση που θα εγκρίνει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή θα είναι η πρόταση προ το Κοινοβούλιο και θα, θα διαβιβαστεί στην Ολομέλεια μετά τη συζήτηση. Και μια πρόκειται για διαδικασία συναπόφαση, θα πρέπει να ζητήσουμε επιβεβαίωση τη εντολή από την Ολομέλεια ε, και μετά να περάσουμε στο τριμερή διάλογο, ενδεχομένω και με την διαδικασία, ε, ανάλογα φυσικά και με τη θέση που θα λάβει το Συμβούλιο. Ω εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω από του κοιόδη να μου πούν τη γνώμη του ε, για το αν συμφωνούν με την προτινόμενη διαδικασία ή αν έχουν κάποιες ενστάσεις ή και σχόλια. Παρακαλώ, ο σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ, τι γνώμη έχει, ο κύριο Φέρμπερ. Σας ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Πρέπει να σας πω ότι είμαστε λίγο απογοητευμένοι ε, και εγώ προσωπικά και η ομάδα μου γιατί άλλαξε λίγο ε, το χρονοδιάγραμμα και μας προκάλεσε κάποια προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Ε, ε, και ε, η πρόεδρος, όχι η σημερινή, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα έπρεπε να μας έχει ενημερώσει πιο πριν έτσι ώστε να προετοιμαστούμε γιατί γίνονται ψηφοφορίες σε πολλές επιτροπές και επομένως δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτά εξ ονόματος ε, της Ιβανα Μάλετιτς ε, μπορώ να πω το εξής. Ε, αυτή η πρόταση ε, αποτελεί τμήμα μιας ε, δέσμης τεσσάρων προτάσεων σχετικά με τους φόρους κατανάλωσης. Η πρόταση αυτή αφορά την ψηφιοποίηση αυτών των φόρων κατανάλωσης για συγκεκριμένα προϊόντα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και πολιτικά μη αμφιλεγόμενο. Ε, και λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμένο χρόνο για συζήτηση ε, στην Επιτροπή που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, συμφωνεί η Σκιώδης με την πρόταση έτσι ώστε να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες έτσι όπως αναφέρονται στον κανόνα 50 εδάφιο 1. Ευχαριστώ πολύ, οι Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Εγώ θα είμαι η Σκιώδης του Σκιώδους γιατί λείπει ο, ο συνάδελφος Και είναι και η πρώτη συνάντησή μας, συνεδρίασή μας στην Επιτροπή ε, Έκονα και εγώ ως συντονίστρια πλέον και όχι ως εκπρόσωπος του Σκιώδους θα ήθελα να ευχηθώ ε, σε όλους ε, τους ε, πολυπληθείς συναδέλφους που βλέπω εδώ καλή χρονιά. Ο κύριος Φανασβλίκα θέλει να πει το εξής. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ε, Θέλω να δουλέψουμε αρμονικά με την εισηγήτρια και τους άλλους ε, σκιώδεις. Ε, εδώ συζητούμε για την περαιτέρω αυτοματοποίηση του συστήματος ε, που αφορά τους φόρους κατανάλωσης και την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκειται σε φόρους κατανάλωσης μέσω απλουστευμένης διαδικασίας που θα επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση αυτών των κινήσεων. Επίσης, δίνεται πλέον η δυνατότητα δυνατότητα αυτοματοποίησης οποιασδήποτε, οποιασδήποτε συστήματος χρησιμοποιείται για τη διακίνηση των αγαθών. Λαμβάνοντα υπόψη ότι η εν λόγω πρόταση δεν ε, προτείνει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή, ε, προτείνουμε ε, να προχωρήσουμε με απλουστευμένη διαδικασία σύμφωνα με τον κανόνα 50 εδάφιο 1 ε, των ε, κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ ε, και προσδοκώ σε καλή συνεργασία όσον αφορά την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Άλντε. Ρεϊμόν Τρεμόσα. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους και από πλευρά Άλντε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, ως συντονιστής και σκιώδης ηγητής πρέπει να σας πω ότι συμφωνούμε με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και με την εισηγήτρια στις προτάσεις της, την κυρία Κέι Σουίμπορν. Συμφωνώ με τους προλαλήσατες συναδέλφους συντονιστές του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και μπορούμε να προχωρήσουμε όπως πρότεινε η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ λέει μόλις Σκοτ Κέιτο από τους Πρασίνους η οποία όμως μου διαβιβάζει ότι σύμφωνοι με τη διαδικασία όπως την περιέγραψα, δεν βλέπω κανέναν από την ενωτική αριστερά. Άλλος κανείς θέλει το λόγο εκτός από τους κοιόδες. Όχι. Η σιωπή προς απάντησή μου. Τη θεωρώ έγκριση της διαδικασίας που σας πρότεινα ως εισηγήτρια για την αποστευμένη διαδικασία για την έκθεση αυτή και θα ζητήσω λοιπόν από τη Γραμματεία να το στείλουμε στην Ολομέλεια αμέσως μετά. Δεν χρειάζεται άλλη συζήτηση. Με γραπτή διαδικασία και προχωρούμε ταχαίως. Ευχαριστώ πολύ. Και τρέχουμε κιόλα. Κανονικά οι ε, ψηφοφορίες άρχιζαν στις 9.30. Που είναι το επόμενο θέμα. Και μετά έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών, ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 19. Ναι, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω μέχρι να έρθει ο εισηγητής. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά να δούμε μήπως έρθει ο κύριος Βαντεν Κέντελαρε. Πώς προφέρεται αυτό το πράγμα. Ο Τόμ, με περιπτώσει, για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Λίγη υπομονή μέχρι να έρθει η τη. Ευχαριστώ. Okay, given that we have the rapporteur here for... Έχει έρθει ο εισηγητής για το επόμενο σημείο της συνημερής διάταξη. Περνάμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Βαντεγκέντελαρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να πέτυχα την προφορά. Τέλεια, Πρόεδρε, το είπατε. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Ε, ακόμα μπορούμε να λέμε χρόνια πολλά και οφείλουμε να λέμε και χρόνια πολλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στι 21 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια ανάλυση τη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο ε, είναι μια πολιτικά ευαίσθητη περίοδο στην Επιτροπή μας, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. Και θα πρέπει να πάρουμε ακριβώς το χρόνο που χρειάζεται για να κάνουμε καλά τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό έκανα ό,τι μπορούσα έτσι ώστε να φέρω το σχέδιο έκθεσής μου ε, ε, πολύ γρήγορα μετά τις 21 Δεκάτου στις 26 Νοεμβρίου. Το έφερα ήδη λίγες μέρες μετά την κατάθεση της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ποιο λόγο, ακριβώς για να έχουμε όσο χρόνο θέλουμε για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε σε βάθος και να διοργανώσουμε όσο γίνεται περισσότερες ε, συνεδριάσεις και οδών εισηγητών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες του παρελθόντος θα πρέπει να διαπιστώσω όμως ότι μόνο τέλη Ιανουαρίου θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και έτσι θα έχουμε λιγότερο χρόνο. Έγιναν πολλές ε, καθυστερήσεις και ολιγορίες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ε, το Συμβούλιο θα το δει ε, το φθινόπωρο. Η ουσία ποια είναι... Ε, διαπιστώνω στην έκθεσή μου ότι ε, υπάρχει μεγάλη γύρανση του πληθυσμού και αυτό είναι τεράστια ε, πρόκληση και χρειάζεται να αντιδράσουμε Αλλά τώρα η συγκυρία δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκή. Βαίνουμε προς το τέλος τη περίοδου. Θα πρέπει να λάβουμε, να λάβουμε δράση, να μην ε, σκεφτόμαστε τι ε, εκλογές, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα βάλουμε συνεχώς. Όσο αυξάνεται, μάλλον στο γυράσκει ο πληθυσμό, αυξάνεται το κόστος για τις συντάξεις και για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Έτσι και αλλιώς είναι πολύ ψηλό το κόστος των συντάξεων και θα αυξηθεί. Θα έχουμε περισσότερες δαπάνες, ε, σας είπα για τις συντάξεις, για την υγεία, για την περίθαλψη και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση. Δεύτερον, όσο γεννάει ο πληθυσμός, είναι λιγότεροι εργαζόμενοι που χρηματοδοτούν τις συντάξεις με τις ε, εργοδοτικές εισφορές, γιατί αυτό είναι αρχή ε, της κοινωνικής ασφάλειας, όπως το γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν με τις εισφορές τους τις συντάξεις των νυν συνταξιούχων, όχι τις δικές τους. Και αυτό ε, είναι κάτι το οποίο γνωρίζει μεγάλη πίεση. Γύρω στο 2070, λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα έχουμε αύξηση κατά 52% στην Ευρωζώνη του όρου συνταξιούχη ε, προς ε, εργαζομένους. Δηλαδή, το 2016 είχαμε τέσσερις εργαζομένους για έναν συνταξιούχο, ε, το 70 θα έχουμε δύο εργαζομένους για έναν συνταξιούχο. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα βλέπουμε σε μια τέτοια διάσταση ε, στο απότερο μέλλον για να προετοιμαστούμε ε, και στα δημόσια οικονομικά μας. Με τρεις τρόπους, το λέω και στην ε, έκθεσή μου, φορολογικά μαξιλαράκια, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και παραγωγικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς το ίδιο προτείνει. Φορολογικά μαξιλαράκια ε, κάποια αποθεματικά για να αντιμετωπίσουμε ε, τη γύρα του πληθυσμού. Σίγουρα, όταν είναι ευγνωκή η συγκυρία, θα πρέπει να βάλουμε τάξη στα πράγματα, όπως σε αυτή την περίοδο. Το πρόβλημα δεν είναι κάποια ποσοστά, είναι σημαντικό στοιχείο για την ε, νομισματική μας ένωση να ακολουθούμε όλους τους κανόνες. Μετά τα φορολογικά έχουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ακριβώς για να μειώσουμε το κόστος της γύρανσης. Γνωρίζουμε ότι ε, είναι λιγότεροι ε, εκείνοι που είναι ενεργοί επαγγελματικά και περισσότεροι συνταξιούχοι. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, τονώσουμε την αγορά. Πιο ευέλικτες αγορές εργασίας, προσαρμοσμένες θα πρέπει ο, ο κόσμος ε, να είναι ευέλικτος, ε, να είναι απασχολήσιμος και να μετακπαιδεύεται. Όχι απλώς ένα δίπλωμα, αλλά και οι δεξιότητες μας ενδιαφέρουν, η διαβίου μάθηση, ε, να μειωθούν τα γραφειοκρατικά και τα διοικητικά εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο κόσμος να μπορεί να εργάζεται περισσότερο, να αποκτά νέες δεξιότητες και προνόμια. Πέρα από αυτά τα δύο, το τρίτο που προτείνω είναι αύξηση της παραγωγικότητας. Θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε ε, συνεχώς για να είναι η φόρος και βιώσιμη η ανάπτυξη στο μέλλον. Και το τονίζω, γιατί καλή είναι η οικονομική ανάπτυξη μεγέθη τη οικονομίας, αλλά βιωσιμότητα μας ενδιαφέρει πιο πολύ. για να εξασφαλίσουμε και τη μελλοντική παραγωγικότητα, αλλά να είναι και παραγωγικές οι επενδύσεις. Θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση στα έξοδα, ε, στις δαπάνες της δημόσιας, ανάμεσα στις τρέχουσες δαπάνες και στην ανάπτυξη. Ε, γιατί έχουμε την ψηφιοποίηση, την έρευνα, την ανάπτυξη. Ε, και εκτός από το φυσικό κεφάλαιο, το οικονομικό δηλαδή, θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Έχω κάνει το σχέδιο της έκθεσης, περιμένω τις συζητήσεις που θα είναι ενδιαφέρον ενδιαφέρουσες, ε, σίγουρα και τα επιχειρήματα των συναδέλφων που θα έχουν και κάποιες διαφωνίες φαντάζομαι, αλλά και θα είναι και επικοδομητικά. Σας ευχαριστούμε. Ακούσαμε τον εισηγητή, θα περάσουμε στους και εισηγητές τώρα. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Περέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το σχέδιο έκθεσης που υπέβαλα. Και σίγουρα θα αποτελέσει τη βάση για μια πολύ ζωηρή συζήτηση και εντατική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η τύση επισκόπηση για την ανάπτυξη και οι κατευθυντήριε γραμμέ και προσανατολισμοί που δίνει για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Συνήθω ξεκινάμε λέγοντα ότι ε, το προτινόμενο σχέδιο έκθεση αποτελεί μια καλή βάση για το έργο μας. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου ε, με το σχέδιο έκθεσης. Δεν είμαι βέβαιος ότι αποτελεί όντως μια καλή αφετηρία για τη συζήτηση, γιατί θα ήθελα να είμαστε βέβαιοι ότι ο εισηγητής είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις πολιτικές ομάδες, προκειμένου να καταλήξουμε σε πολιτικούς συμβιβασμούς. Βέβαια, δεν μας ευνηδιάζει αυτή η διάσταση απόψεων που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, οικονομική, για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, αλλά συνήθως ξεπερνούμε τις πολιτικές μας διαφορές προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Βέβαια, η διατύπωση του σχεδίου έκθεση με προβληματίζει για το κατά πόσο είναι δυνατή μια τέτοια υπέρβαση των διαφορών. Και δεν είμαι βέβαιο πόσο ε, διαλλακτικό και πόσο πρόθυμο θα είναι για συμβασμού ο εισηγητή, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Και σίγουρα η ομάδα μου έχει την πολιτική βούληση και προθυμία για συζήτηση και ανέβρεση συμβαστικών προτάσεων. Βέβαια, διαβλέπουμε αρκετές πολιτικές δυσκολίες στη διαδικασία. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι για την πολιτική μου παράταξη η ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται αρκετά ισορροπημένη. Και θα θέλαμε και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποστηρίζει την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτή διατυπώνεται στην ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη, κάτι που δεν ισχύει με το συγκεκριμένο σχέδιο έκθεσης του κ. άρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα, μας υπέβαλε και πρότεινε τρεις προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η υψηλή ποιότητα επενδύσει και ιδιωτικέ και δημόσιε. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι οι μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί όχι μόνο η παραγωγικότητα, αλλά και η συμπερίληψη, η συμμετοχή και η ποιότητα δημοσιονομική και επίσης μακροοικονομική σταθερότητα και ε, υγιή δημόσια οικονομικά. Ε, είναι διαφορετικές όμως οι προτεραιότητες του εισηγητού. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η δημιουργία δημοσιονομικών αποθεμάτων. Πολύ διαφορετική προσέγγιση και προτεραιότητα από αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργία δημοσιονομικών αποθεμάτων, ε, συγκράτηση του μισθολογικού κόστους. Αυτό δεν είναι πρόβλημα βέβαια. Αλλά το πρόβλημα είναι εκεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ω προτεραιότητα την δημιουργία μακροοικονομικής σταθερότητας, γιατί η δημοσιονομική πειθαρχία είναι ένα στοιχείο αυτή τη μακροοικονομική σταθερότητα, ο εισηγητή προτείνει κάποια δημοσιονομικά μαξιλαράκια, κάποια δημοσιονομικά αποθέματα και διαγράφει πλήρω κάποια μνήμα τη μεταρρύθμιση οικονομική και Νομισματικής Ένωσης, που είναι απαραίτητο στοιχείο τη δημιουργία μακροοικονομικής σταθερότητας. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του εισηγητού, αλλά έχουμε πρόβλημα και με το περιεχόμενο, με την ίδια την προσέγγιση του εισηγητού στι προτεραιότητες που διατυπώνει. Και η πρώτη προτεραιότητα, όπως σα είπα, είναι αυτή για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Το ίδιο ισχύει και με την προτεραιότητα του εισηγητού, ε, με την προτεραιότητα μάλλον για τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επενδύσεις υψηλής ποιότητας στην έρευνα, την παιδεία, τις δεξιότητες, τις υποδομές. Ενώ η συγητής αναφέρεται κυρίως στις επενδύσεις για την παραγωγικότητα, για το παραγωγικό σκέλος της οικονομίας. Μια, δηλαδή, πρόταση χειρότερη από αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ο εισηγητής επιμένει στην ιδέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μείωση του δημοσιονομικού κόστους και κάποιες ε, δημόσιες παρεμβάσεις για τις ε, ε, συντάξεις και η πρόθεση μιας ελαστικής αγοράς εργασίας. Και δεν λαμβάνει υπόψη την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ευρεία συμμετοχή και αποφυγή αποκλεισμών. Και αυτό πραγματικά μα δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα με τις προτεραιότητε του εισηγητού, έχουμε πρόβλημα με την προσέγγιση που υθετεί για τις διάφορες προτεραιότητε και θα θέλαμε μια έκθεση που θα ευθυγραμμίζεται πολύ περισσότερο με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πιστεύω ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση θα καταλήξουμε σε, πολιτικές, σε πολιτικούς συμβιβασμούς. Αλλά θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι όντως είναι πρόθυμος να αναζητήσει πολιτικούς συμβιβασμούς ε, ο εισηγητής μας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ τώρα. Ο σκιώδης ηγητής Ρόμπερτ Σίλα απουσιάζει και ο συντονίστρια θα διαβάσω τι σημειώσει του. Ε, ζητώντα εκ μέρου του συγγνώμη για την απουσία του. Ο κύριο Τζίλη, λοιπόν, ευχαριστεί τον εισηγητή για την καλή του προσπάθεια και χαιρετίζει την έκθεση του. Θεωρεί ότι ο εισηγητή πολύ σωστά εντόπισε τα περισσότερα ζητήματα και τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωζώνη και το Σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθησε να υιοθετήσει μια ισορροπημένη άποψη ο εσκόδης του ECR θεωρεί ότι θα έχουμε επικοδομητική περαιτέρω συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε, πολύ σωστά τονίζεται η ανάγκη για δημοσιονομικά αποθέματα. Δεδομένων όμω των προκλήσεων αλλά και τη γύρανση του πληθυσμού τη Ευρώπη, είναι σημαντικό να έχουμε και αύξηση τη παραγωγικότητα. Επίση, ο σχεδόν συγκεκριτή μα πιστεύει ότι εδώ υπολοιπο... υστερούμε κάπω. Και χωρί αύξηση τη παραγωγικότητα δεν θα έχουμε πραγματικά δημοσιονομικά πλεονάσματα ή δεν αρκούν αυτά. Επίσης, περαιτέρω μείωση της ανεργίας και ακόμη πιο σημαντικό της υποαπασχόλησης και η μείωση της ε, μείωσης ε, του, της ε, ηλεκτρονικής, της οικονομίας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Επίσης, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ε, όντως το δημοσιονομικό χρέος είναι πάνω το 60% στα περισσότερα κράτη-μέλη, αλλά έχουμε και σημαντικά ελλείμματα. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να δαχτυλοδεικνυουμε μονο μόνο κάποια κράτη-μέλη. Η Ιταλία είναι ακραίο παράδειγμα, αλλά άλλα τέσσερα κράτη-μέλη στο 2019 υπέβαλαν δημοσιονομικά σχέδια που ε, να έχουν τον κίνδυνο τη μη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Επίση, χαιρετίζουμε το γεγονό ότι ο εισηγητή αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν μόνο ε, αρνητικέ αλλά και θετικέ ανισορροπίε, όπω κάποια πλεονάσματα δημοσιονομικά κάποιων κρατών μέλων. Και αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ο κύριος Ζήλε θεωρεί ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήδη περνάμε σε ένα πολύ κρίσιμο κλίμα περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης. Δεν θέλει να είναι απεσιόδοξο, αλλά προσεκτικός ο κύριος Ζήλε ε, κατά τις άποψη ότι έχουμε ξεπεράσει τα πιο δύσκολα, γιατί και μπροστά μας έχουμε αντικσότητες. Ίσως από αυτήν την άποψη παρά είναι αισιόδοξη η έκθεση του εισηγητού. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Ζηλετή χαιρετίζει και προσβλέπει σε πολύ επικοδομητική συνεργασία. Εξ ονόματος ε, της ε, Άλντε δεν έχουμε εκπρόσωπο εδώ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, έχουμε. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λέω ο κύριος ε, και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή κύριο Τόμ Βαντεν Κίντελαρ γιατί η έκθεσή του αποτελεί μια καλή βάση προς συζήτηση σε γενικές γραμμές μπορώ να συμφωνήσω με την κατεύθυνση που παίρνει ε, η έκθεση αυτή εστιάζει σε μελλοντικέ προκλήσεις όπως α πούμε ε, το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί γιατί είναι θεμελιώδο σημασία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί περισσότερο η δύναμη της νεολαίας στην ενιαία αγορά. Ε, επίσης το θέμα των ε, δημοσιονομικών αποθεμάτων, των buffers, είναι κάτι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να ξεπεραστούν κάποια δημόσια χρέη και μεγάλα ελλείμματα προβλήματα σε ορισμένες χώρες μέλη. Βλέπουμε επίσης ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεωθεί να παρέμβει θα πρέπει να ενδυναμωθεί κατά κάποιο τρόπο το κείμενο, ας πούμε ζητώντας ανάλυση ε, βιωσιμότητας ε, για όλες ε, τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις να ζητηθεί αυτό από την Κομισιόν. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό μέσω των τροπολογιών μου. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την κατεύθυνση του εισηγητού και όσον αφορά τις επενδύσεις και την αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά την Νομισματική ε, Ένωση και τι ε, δράσεις θα πρέπει να αναλυθούν ε, εν τέλει. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να δείξουν επιμέλεια και επομένως θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί καλό συντονισμός μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Κομισιόν. Όπως ήδη είπα, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες με στόχο τη βελτίωση του κειμένου, ωστόσο σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και είμαι βέβαιος ότι εν τέλει θα επιτύχουμε ένα πολύ καλό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή ε, και οπωσδήποτε προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους κοιόδης. Άκουσα πολύ προσεκτικά και τα όσα είπε ο Πέδρος Σίλβα Περέιρα. Ξέρουμε ήδη κάποια στοιχεία σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί ε, και είμαι ε, σίγουρος ότι θα μπορέσουμε από κοινού και μέσω συζήτησης και διαλόγου να βρούμε μια ισορροπημένη λύση σε όλα τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόρβαλτς. Δεν βλέπω κάποιον από τους πράσινους. Είχαμε τον Σκιώδια, ο οποίος εξυφανίστη μυστηριωδώς. Θα δούμε εάν ε, επανέλθει να του δώσουμε το λόγο. Επίσης από την Ενωτική Αριστερά, Γκουέ δεν βλέπω κάποιον. Ούτε από την EFTD. Ούτε και την κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ βλέπω από το ΙΕΝΕΦ. E Άρα ε, περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Thank you very much and uh, thanks to the ο κύριος ε, Χοκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την καλή του ε, εργασία. Ε, είδα ότι ο Σκιώδης ε, των ε, σοσιαλιστών ήταν αρκετά ικανοποιημένος. Μην ζητάμε και υπερβολικά πράγματα. Φαίνεται να υποστηρίζει την κεντρική κατεύθυνση της έκθεσης και αυτό μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή συζήτηση για, τα, για μελλοντική συζήτηση. Μην κοιτάτε έτσι τόσο κακύποπτα. Το σημαντικό πάντως εδώ είναι να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά θεμελιώδους σημασία. Είναι υπερβολικά πολλά τα κράτη-μέλη τα οποία υστερούν όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη ε, δυνητικής ανάπτυξης ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και της οικονομίας των μεμονωμένων μελών. Ε, μιλάμε για προβλήματα στην ευρωπαϊκή οικονομία και εγώ το λέω και το ξαναλέω, επανέρχομαι σε αυτό πολλές φορές. Συζητούμε πάντα τον μέσο όρο ανάπτυξης και λέω συχνά ότι εάν ας πούμε έχεις ε, το κεφάλι σου μέσα σε ένα ψυγείο και τα πόδια σου στο φούρνο μπορείς να βρεις μια μέση θερμοκρασία η οποία όμως δεν θα αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ασθενέστερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα να ε, προωθηθούν και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Προβληματίζομαι λοιπόν όταν ε, οι σοσιαλιστές ε, φίλοι μας ε, στεναρά αντιστέκονται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί όμως εδώ είναι το πρόβλημα και αυτό υπονομεύει τα δημόσια οικονομικά και με αυτόν τον τρόπο καθαρά θα χάσουμε απέναντι σε άλλα μέρη του, της υφηλίου λόγω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας η οποία κινείται γρήγορα και εν πάση ε, περιπτώσει κινείται ταχύτερα σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη κούρσα ε, και δεν μιλάμε για κούρσα προς τα κάτω, είναι πάντα κούρσα προς τα πάνω, προς την κορυφή. Και ακριβώς γι' αυτό χρειάζονται οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Και εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία ε, και οι σοσιαλιστές, γιατί διαφορετικά μόνο προβλήματα θα έχουμε μπροστά μας, μόνο προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε ότι ολοκληρώνεται, ε, κλείνει προς τα κάτω ο οικονομικός ε, κύκλος. Αυτοί οι οποίοι ε, ε, δεν δέχονται τις με, ε, μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανοίγουν ολιστηρό μονοπάτι προς την ανεργία και τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Περβάνς Μπερές, ευχαριστώ πολύ. Ζωντανή η συζήτηση και είναι πολύ καλό αυτό. Στόχος δεν είναι να δούμε αν η ευρωπαϊκή οικονομία πάει καλά, αλλά ε, η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι ε, στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά που είπε ο κύριος Σόκμαρτ είναι ενδιαφέροντα, αλλά πρέπει να σας πω ποια είναι η θέση της σοσιαλιστικής ομάδας, έτσι όπως εξεφράστη από τον Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ε, λέτε αγαπητέ συνάδελφε ότι έχει, έκανε μια ε, γενική θετική εκτίμηση. Ναι, αλλά γενική θετική εκτίμηση της ε, πρότασης της Κομισιόν και όπου και πρέπει να πούμε όμως ότι η, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων για τον επόμενο χρόνο μέσω της επισκόπησης είναι πάρα πολύ σαφής. Όμως αυτή η διαδικασία όχι μόνο δεν ε, την ενστερνίζεται ο, ο, ο εισηγητής, αλλά την αντιστρέφει. Και ξεκινώντας από τα ε, διδάγματα της προηγούμενης θητείας ε, και ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο πρόεδρος Γιούγκερ έλεγε ότι η ποιότητα των επενδύσεων είναι το πιο σημαντικό, ο εισηγητής όχι μόνο δεν λαμβάνει την τρίτη προτεραιότητα υπόψη που λέει «Ensuring macroeconomic stability», υγιή, δημόσια οικονομικά και λοιπά Αλλά την ε, μεταφέρει διαφορετικά λέγοντας ότι χρειάζονται μεγαλύτερα δημοσιονομικά αποθέματα. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια ερμηνεία η οποία πολύ διαφέρει και από τις προτεραιότητες ε, της Κομισιόν αλλά και από τη διατύπωση των προτεραιοτήτων. Και να προσθέσω και άλλες δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, η ιδέα του εισηγητή ότι από τη μία πλευρά είναι αυτοί που θέλουν να σεβαστούν τους κανόνες και από την άλλη πλευρά αυτοί που θέλουν εντελώς να αλλάξουν εντελώς τους κανόνες. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κανόνες που να είναι συνεκτικοί, να έχουν μια λογική σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει. Θέλουμε ευρωπαϊκή οικονομία με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ωραία, αλλά η εμπειρία μας δείχνει ότι οι, ισχύουν, οι ισχύοντες κανόνες είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι, δεν επιτρέπουν την ε, ε, σωστή τους ε, εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και Επίσης θα ήθελα για μια τελευταία φορά ε, να σπάσω αυτό το απόστημα, το έκανε και ο Σκιώδησε. οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες είναι υπέρμαχοι της ε, διαφορετικής ε, μεταρρύθμισης, αλλά όχι της τυφλής και χωρίς κατεύθυνση ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναρχίσουμε από το μηδέν. Και αυτό που διαπιστώνουμε και ο εισηγητής το είπε είναι ότι ενώ η Κομισιόν έχετε με συγκεκριμένες προτάσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που μας φαίνονται θεμητές, ε, τις απορρίπτει ο εισηγητής. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ε, τον κόσμο έτσι ώστε να ενισχύσει αυτό που εσφαλμένα ενδεχομένως ονομάζουμε ε, ανθρώπινο κεφάλαιο. Ε, ε, εν πάση περιπτώσει, τα λέμε και τα ξαναλέμε τα ίδια πράγματα, ε, αλλά ξέρουμε ότι εάν θέλουμε να ενισχύσουμε κάποιες ε, ε, μεταρρυθμίσεις ε, θα πρέπει ενδεχομένως να μιλήσουμε πρώτα για σύγκληση έτσι ώστε να μην ενεφερόμαστε μονάχα στα ελλείμματα κάποιων χωρών αλλά και στα πλεονάσματα κάποιων άλλων χωρών. Αυτά ήθελα να πω και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά δεν είμαστε και πολλοί σήμερα εδώ, οπότε θεώρησα ότι μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Μπέρες. Ελπίζω όμω να μην καθυστερήσουμε τι ψηφοφορίες που προβλέπονται για αργότερα. Ο εισηγητή τη Επιτροπή των Περιφερειών για το θέμα αυτό ζήτησε το λόγο. Κύριο Γιόγκμαν, ε, έχετε λίγα λεπτά, κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που δίνετε το λόγο και στην Επιτροπή των Περιφερειών και την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Συνήθω το αντίστροφο συμβαίνει. Εσεί, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έρχεστε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Τώρα συνέβη το αντίθετο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Στη νέα της επισκόπηση για την ανάπτυξη έχουμε μια πολύ καλέ ειδήσει. Καταρχήν, επικεντρώνονται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν ε, για τι επενδύσει που χρειάζονται σε τομεακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παρόλο που η περιφερειακή διάσταση παρά είναι μικρή ακόμη. Και για πρώτη φορά επίσης αναφέρονται οι εδαφικές ε, διαφορές, κάτι που ζητούσαμε έντονα τα τελευταία χρόνια στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και μάλιστα οι ειδικέ ένα αναχώρα και οι εκθέσει αναχώρα από εδώ και πέρα θα λαμβάνονται υπόψη στη, στον προγραμματισμό τη πολιτική συνοχή. Αλλά δεν είναι ο μόνο λόγο που το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, ενδιαφέρει όλο και περισσότερο και έχει μεγαλύτερη σημασία σε εθνικό επίπεδο. Τα νέα προγράμματα στήριξης των μεταρρυθμίσεων θα δώσουν ενάυσματα για την εκπλήρωση των μεταρρυθμιστικών υποχρεώσεων που εντοπίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Οπότε είναι ακόμη πιο σημαντικό να ασχοληθούμε με μερικά κέρια σημεία. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, αλλά σε ποιε ακριβώ διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Δεύτερον, πώ μπορούμε ελαστικά να αντιμετωπίσουμε τα διαφοροποιημένα προβλήματα που έχουν οι αστικές σε σχέση με τις ε, ε, αγροτικές περιοχές και περιφέρειες. Επίσης, να μην μείνουν πίσω οι, οι περιφερειακές, ε, περιφερειακά εδάφη σε σχέση με τα κεντρικά. Πώς θα προωθήσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, γιατί εκεί είχαμε αρκετά προβληματική κατάσταση μέχρι στιγμής. Επίσης, πώς θα αποφύγουμε παραβάσεις αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Γιατί με τέτοιες παραβιάσεις, ε, μάλλον θα υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις, αν δεν έχουμε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση με λήψη υπόψη τη διαφορά των περιφερειών στην πολιτική συνοχή. Και ιδιαίτερα σε περιπτώσει που δεν έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μερικέ φορέ έχουμε και ανύπαρκτη κοινωτική αρμοδιότητα. Η άποψή μας είναι ότι τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να λυθούν αν όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης συνεργάζονται στενά για το σχεδιασμό και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και παρά κάποιες θετικές πρακτικές, αυτή τέτοια συνεργασία δεν υπάρχει. Το 2017 μάλιστα προτείναμε ένα διεντολογικό κώδικα, κώδικα συμπεριφοράς για τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Και μάλιστα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του Οκτωβρίου 2016 στενίστηκε αυτή την άποψη. Δυστυχώς ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντέδρασε θετικά, δεν εισάκουσε την ε, πρότασή μας για ένα διοντολογικό κώδικα. Και αυτό πραγματικά μας οδήγησε ένα παράδοξο, γιατί οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στα πλαίσια της ε, περιφερειακής πολιτικής ε, στηρίζονται στο διδατολογικό κώδικα της αρχής της εταιρικής σχέσης που εξασφαλίζει συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων. Αλλά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν υπάρχει νομική βάση για την ανάμεξη και συμμετοχή των δήμων και περιφερειών. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευθυγραμμίσει την πολιτική συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και αυτό το παράδοξο δεν προβληματίζει μόνο τους δήμους και τις περιφέρειες. Η Ρουμανική Προεδρία ζήτησε από την Επιτροπή των Περιφερειών να συντάξει σχετική γνωμοδότηση. Το τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό σημείο μου είναι ότι το Ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν είναι αυτός σκοπός. Μέχρι στιγμή, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η πολιτική συνοχή ευθυγραμμίζονται με του στόχου ε, τη ε, στρατηγική για το 2020 για την Ευρώπη, που φτάνει στο τέλο τη. Χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για να μπορούν καλύτερα οι ενδιαφερόμενοι και οι δημόσιες αρχές να ανταλλάξουν τις απόψεις για τις προοπτικές που προτιμούν. Επίσης θα πρέπει να δοθούν κάποια ανταλλάγματα ε, και να βρούμε μια εξισορρόπηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της μακροοικονομικής σταθερότητας. Ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά, ώστε να εξασφαλίσουμε το νέο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να πραγματοποιήσει ένα ποιοτικό άλμα σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνης γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία και την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιόγκμαν. Ο εισηγητής τώρα για να κλείσει και να συνοψίσει. Κύριε Βαντοκεντελάρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Πρώτον, να τιμήσουμε και την Ευρωπαϊκή, την ε, Επιτροπή των Περιφερειών για την παρουσία της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει και στις 21 Ιανουαρίου ε, θα τους παρουσιάσω την ε, έκθεσή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει και η Επιτροπή των Περιφερειών ε, πρέπει να συμμετέχουν όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης για να μπορούν να εφαρμοστούν οι συστάσεις ανά χώρα αποτελεσματικά. Συμφωνώ απολύτως για την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή. Αν θέλουμε να κάνουμε προόδους είναι κρίσιμος ο ρόλος τους. Και τα εθνικά κοινοβούλια και τα περιφερειακά κοινοβούλια αλλά και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ περισσότερο υπόψη στη συζήτηση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Εκείνοι γνωρίζουν τις ανάγκες ε, κυρίως για τις μεταρρυθμίσεις και τις τις επενδύσεις. Ε, εκτός αυτού ε, είναι σωστό ότι θα πρέπει να έχουμε ε, θεσμική ικανότητα και διοικητική ικανότητα. Και συμφωνώ με τον κώδικα δεοντολογίας που προτείνει η Επιτροπή των Περιφερειών. Κάθε επίπεδο διακυβέρνησης έχει τις προτεραιότητές του και θα πρέπει να τολμούμε να επιλέγουμε ε, το σωστό επίπεδο κάθε φορά, την κάθε προτεραιότητα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούσαμε σήμερα τη φωνή τη Επιτροπή των Περιφερειών. Έρχομαι τώρα στου συναδέλφου μου και οδησηγητές. του ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ για τη θετική και επικοδομητική κριτική που εκφράζουν να πω ε, μερικά πράγματα προς τους ε, σοσιαλιστές ε, συναδέλφους για τα επικριτικά σχόλια. Κοιτάξτε, σε μια τέτοια έκθεση είναι περιορισμένος ο χώρος, ακόμα και οι χαρακτήρες και οι λέξεις που χωράνε και πρέπει να επιλέγω. Βεβαίως να πούμε ό,τι θέλετε για τις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, να συζητήσουμε και τη σημασία των ποιοτικών επενδύσεων και τη θεσμική και διοικητική ικανότητα χωρίς αποκλεισμούς και τη συμπερίληψη. βεβαίω, κυρία ε, ε, ε, είμαι πρόθυμος να μιλήσω για απλούστευση. Αν είχατε διαβάσει την έκθεση μου θα τα είχατε δει όλα αυτά. Δεν μιλάω για τις χώρες μόνο με ελλείμματα αλλά και για τις χώρες με πλονέασματα. Αν μελετήσατε την έκθεση θα είδατε ότι στην παράγραφο 6 λέγει ότι χαίρομαι κυρίως για τις τρεις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είστε κι εσείς ως ομάδα πρόθυμοι να τις υιοθετήσετε. Αυτό λέω για τις μελλοντικέ συζητήσεις μας. Πώς θα γινόταν διαφορετικά. Θυμάμαι μια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε το συνάδελφο ε, Ιγκ Μπαγιέ, αλλά δεν ε, το στηρίζει πάντα αυτό η ομάδα σας. Το πλαίσιο λοιπόν είναι σαφέστατο. Πρέπει όμως να περιμένουμε και ε, από ένα ε, εισηγητή να κάνει συμβιβασμούς. Εγώ είμαι Βέλγος. Εκτός από τις τηγανιτές πατάτες εδώ και τη σοκολάτα, έχουμε παράδοση εμείς και στους συμβιβασμούς. Είμαστε πάντα ε, στη διάθεσή σας για τους συμβιβασμούς. Ε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Περέιρα, εσείς είστε πρόθυμοι για συμβιβασμούς. Γιατί περισσότερο από ποτέ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και ενώπιση των ευρωεκλογών που οι συμβιβασμοί δεν είναι για να έχουμε βγάλει μια ωραία φωτογραφία στο τέλος της έκθεσης, αλλά για να έχουμε εξασφαλίσει τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον εισηγητή και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Θα σας δώσω τώρα για να τελειώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό, το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, Προθεσμία για τις τροπολογίες 17 Ιανουαρίου του 2019. Μελέτη των τροπολογιών, εξέταση των τροπολογιών 25 Δευτέρου του 2019. Ενδεχομένως όμως ε, μπορεί να γίνει και 26 αυτή η ημερομηνία, 26 Δευτέρου. Η ψηφοφορία ε, στην πρώτη ολομέλεια του ε, Μαρτίου. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τη συμβολή σας στη συζήτηση αυτή. Και μια και έχουμε τον χρόνο, θα μπορούσαμε να πάρουμε την επόμενη έκθεση, αλλά ο εισηγητής ε, ζήτησε συγνώμη ε, για την απουσία του και ζητά από τον κύριο Φαντελάρε μήπως μπορεί να παρουσιάσει το θέμα. Δεν ξέρω και αν και οι εισηγητές είναι εδώ. Is he coming or are you doing it? Okay. And I'm doing it on behalf of Mr. and therefore I think we can... Ωραία, εγώ θα μιλήσω για το εξονόμητος του κυρίου Ζήλε. Δεν ξέρω αν ξέρετε αν ο κύριος Κόφοντ θα έρθει. Θα δούμε, θα δούμε. Κύριε Βάντεν Κάντελάρε, να μιλήσετε για το επόμενο θέμα, εισαγωγή αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματο ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών. Ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Βαν Καντελάρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, έλαβα μία πάρα πολύ ε, ε, λεπτομερή εισήγηση από τον κύριο Μαρτουσέλο. Πρώτα απ' όλα με ευχαριστεί γιατί τον εκπροσωπώ και, γιατί, και ζητά συγγνώμη γιατί δεν είναι εδώ. Ε, ήταν σαφές ε, ότι όλα τα μέτρα ε, για το οριστικό σύστημα ΦΠΑ είναι κάτι που χρειάζεται η Ευρώπη και το χρειάζεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό υπάρχει ένα καινούριο πλαίσιο το οποίο θέλουμε να αντικαταστήσει το παλαιό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε βελτίωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά τα ενδιαφέροντα αριθμητικά στοιχεία τα οποία υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι σημαντικό και για τους πολίτες ε, ε, μια και ε, σημαίνει ότι εφογκραζόμαστε τις ανάγκες και τις ανάγκες της κοινωνία. Το νέο σύστημα το οποίο έχει υποβληθεί ε, βάσει της ε, νέας ε, οδηγίας έχει αρκετούς στόχους μεταξύ των οποίων την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι αρκετά εύκολο εάν λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να χτυπηθεί αρκετά εύκολα. Επίσης μπορεί να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα των αφανών εμπορευομένων. Με το θέμα αυτό μιλάμε πλέον ε, όχι για ε, διακοινωτική διακίνηση αγαθών αλλά ε, για μετακίνηση απλή αγαθών εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μιλάμε εδώ για κέρδος το οποίο να φτάσει, μπορεί να φτάσει στα 43 δις ευρώ. Ε, ο κύριος ε, Μαρτουσέλο ε, θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιες ιδέες οι οποίες είναι σημαντικές και έχουν προέλθει από άλλες, από άλλες πολιτικές ομάδες όπως η Άλντε ας πούμε η οποία μέσω κάποιων μικρών τροπολογιών μπορεί να συμφωνήσει με την έκθεση. Μιλάμε εδώ για τον ΦΠΑ λόγω του οποίου μπορεί να υπάρξει απώλεια 50 δις κάθε χρόνο. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρξει ένα πολύ ε, γλωσσό ε, ε, πόρταλ το οποίο να βοηθά τους εμπορευμένους. Επίσης είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα του υποκείμενου σε φόρο και την, το χρονοδιάγραμμα. Οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν στην προκείμενη περίπτωση δεν χρειάζεται να έχουμε συνεδριάσεις ε, για την συζήτηση των τροπολογιών ε, ούτε για εξέβρεση συμβιβαστικών τροπολογιών. Επίσης να σας πω ότι ο κύριος Ματρουσέλο θα είναι πάντα στη διάθεση των σκιωδών καθώς επίσης ε, και το γραφείο του. Ε, επίσης, ε, μια και ο κύριος ε, Μαρτουσέλο δεν είναι σήμερα παρόν, μπορείτε να του στείλετε μέσω ηλεκτρονικού θερμίου όλες ε, τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Όλο αναπληρωτές έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ και η κυρία Μπέρες εκ μέρους του κύριου Κοφότ. Ευχαριστώ. Όντω, έτσι ξεκινάω το 2019 με όλο οι σκιώδη στου σκιώδου. Εκ μέρου του κύριου Κοφόντ, θα ήθελα Καταρχήν ε, να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του και να σας πω ότι η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών χαιρετίζει θερμότατα τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει για την έκθεση αυτή που περιστρέφονται γύρω από το άρθρο 13 για τον ορισμό του καθεστώτος αυτού του CTP και θέλουμε ένα σαφέστερο ορισμό και μάλιστα ως ε, ε, εισηγητής για την ε, εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων, ο κύριος Κοφότ χαίρεται που υπάρχει θερμή υποστήριξη για διαφάνεια ό,τι αφορά την χορήγηση αυτού του καθεστώτος του CTP και οι σοσιαλιστές θεωρούν πολύ σημαντικό ότι και το Συμβούλιο σέβεται τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το καθεστώς αυτό που θα είναι τρόπος να παταχθεί η διασυνοριακή φορολογική απάτη του ΦΠΑ που έχει εκτιμηθεί ως 41 δισεκατομμύρια ετησίως αυτή η φοροδιαφύγη. Σε ό,τι αφορά την πιθανή εναλλακτική λύση για το καθεστώς του CTP, είναι σημαντικό να ε, υιοθετήσουμε μια σημαντική θέση. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αντιστάθμισης, ε, οι σοσιαλιστές ε, θα ήθελαν καλύτερη περιγραφή του, της μορφής που θα έχει τέτοιος μηχανισμός αντιστάθμισης και καταθέσαμε και σχετικές τροπολογίες σε σχέση με το έργο και της Επιτροπής Tax 3. Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια θέλαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και να μας πει τι προβλέπει για την έκβαση σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ. Και ευχαριστούμε και τον εισηγητή αλλά και τους υπόλοιπους και εισηγητές, για την επικοδομητική του συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Μπέρε. Θα ήθελα εδώ να εκπροσωπήσω τον σκιώδη εισηγητή του ΙΣΙΑΡ, τον κύριο Τζίλε, που όπως σας είπα, στα συγγνώμη για την ε, απουσία του σήμερα γιατί είχε άλλε ανελημμένες υποχρεώσει. Συμφωνεί και ο κύριο Ζήλε ότι η διασυνοριακή ε, απάτη του ΦΠΑ είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα των κρατών μελών και σίγουρα είναι ραγδαία εξέλιξη οικονομίας και η φορεσπρακτική ικανότητα για το ΦΠΑ δεν ε, ακολουθεί. Ε, και έχει μειωθεί βέβαια το χάσμα σε σχέση με το 2015, ε, που ήταν 12,5% αλλά σε πολλές χώρες εξακολουθεί να είναι 20% και πάνω. Και μάλιστα ε, ένα μεγάλο τμήμα αφορά την απάτη του ΦΠΑ, τη φοροδιαφύγη του ΦΠΑ. θα πρέπει να βελτιωθεί η διασυνοριακή φορή πρακτική ικανότητα του ΦΠΑ. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2012 μάλλον πολιτικά δεν είναι εφικτά για την ίσπραξη στη χώρα προέλευσης. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποιε εμβολίε και για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εφαρμόζει σύστημα ΦΠΑ με βάση την αρχή του προορισμού. Στην ουσία θα υπάρξουν δύο παράλληλα συστήματα για τι συναλλαγέ όταν ε, ο αγοραστής είναι φερέγγιος φορολογούμενος ε, και σε ό,τι αφορά το πιστοποιημένο υποκείμενο στο φόρο, ε, ο κύριος Ζήλε θεωρεί ότι χρειάζεται μείωση της γραφειοκρατίας και μείωση του, του κόστου συμμόρφωσης ε, με τις διατάξεις του ΦΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόθεση είναι καλή και αγαθή, αλλά το καθεστώς του πιστοποιημένου υποκείμενου στο φόρο δεν θα είναι ευνοϊκό για τι επιχειρήσει. για αυτέ που δεν θεωρούνται φερέγγι φορολογούμενοι. Ιδιαίτερα όταν δεν θα εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς κάποιες επιχειρήσεις. Οπότε το καθεστώς ETP ε θα πρέπει να περιοριστεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ίσως κάποιοι ανέντιμοι θα χρησιμοποιήσουν το καθεστώ CTP για να συνεχίσουν τη δουλειά του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό υπογράμμισαν και οι ακαδημαϊκοί αλλά και οι εμπειρογνώμονε. Και μάλιστα ε, ο κύριο Ζήλε ε, συμμερίζεται τι αμφιβολίε των κρατών μελών ότι τα κριτήρια εφαρμογή του CTP είναι πολύ αόριστα και ίσω οδηγήσουν σε διαφορετική ερμηνεία από τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, ο σκιώδη ε, του ECR είναι αισιόδοξο ότι υπάρχει δυνατότητα ανέβρεση συμβαστική λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπει σε επικοδομητική συζήτηση. Δεν βλέπω κανένα από του φιλελεύθερου όμω να ζητά το λόγο, οπότε περνάω στους πράσινους, στην κυρία Μόλι Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ, Κέι. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ότι θέλουμε ένα ενοποιημένο σύστημα ΦΠΑ και οι πράσινοι χαιρετίζουν τον καλύτερο συντονισμό των φορολογικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το είδαμε στις διάφορες επιτροπές τάξη τι πρόβλημα δημιουργείται όταν δεν έχουμε ενοποιημένο σύστημα φορολογίας γιατί αξιοποιούνται τα παραθυράκια του και οι κερκόπορτές του από τους ανέντιμους θέλουμε, χαιρετίζουμε τη μετάβαση από ένα περίπλοκο και μεταβατικό μακροχρόνιο μεταβατικό σύστημα σε ένα οριστικό επιτέλους σύστημα ΦΠΑ. Η έκθεση του κ. Μαρτουσέλο αναγνωρίζει ότι το ισχύον καθεστώς ΦΠΑ έχει πολλές αδυναμίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη φορολογία στην προέλευση και το υψηλό κόστος συμμόρφωσης και αφήνει πολλά παραθυράκια για απάτη. Στην τροπολογία 26 ε, λέμε ότι θα πρέπει... Ε, ο να, και το καθεστώς αυτό να επιτρέπει την καλύτερη ανέβρεση των ανέντιμων ε, ε, φορολογούμενων που δημιουργεί κατά κάθε χρόνο φοροδιαφύγει ύψου 50 δισεκατομμύριων και το, μάλιστα το 2016 ήταν 147 δισεκατομμύρια με βάση εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εισαγωγή του πιστοποιημένου υποκείμενου στο φόρο για τις ε, φερέγγε επιχειρήσεις που κάνουν ενθουσιακές συναλλαγές, η, ο ΦΠΑ ε, καταβάλλεται στο χώρο, στη χώρα προορισμού. Αυτό είναι καλό γιατί πλουστεύεται η κατάσταση για τους ε, φερέγγιους φορολογούμενους, αυτούς που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιοι. Και παρόλο που επί της αρχής είμαστε ε, υπέρ της αρχής, στην ουσία ίσως δημιουργηθούν κάποια παραθυράκια και στις τροπολογίες 47 ε, ε, και 48 ε, μιλούμε για τους όρους υπό τους οποίους θα δοθεί αυτό το καθεστώς του πιστοποιημένο υποκείμενο στο φόρο και την ανάγκη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών. Προσβλέπουμε πάντω σε πολύ καρποφόρε συζητήσει και με του υπόλοιπου και οδησίγητε. Ευχαριστούμε κυρία Σκοτ Κέιτο. Δεν βλέπω κανένα και εκπρόσωπο τη ΚΟΕ. Για το EFTD κανεί. Κανεί, αλλά ούτε και από το ENF υπάρχει εκπρόσωπο. Οπότε επειδή έφυγε και ο αναπληρωτή ε, ε, εισηγητή, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει να πει κάτι. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Um, uh, Ετέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με το που βρίσκεται η κατάσταση στο Συμβούλιο των συζητήσεων. Μέχρι τώρα έχει συνεδριάσει έξι φορές η αρμόδια ομάδα εργασία σε τεχνικό επίπεδο. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στις συζητήσεις αυτές η πρόταση πρέπει να αλλάξει γύρω στις 200 διατάξεις στην οδηγία για το ΦΠΑ. Αυτές οι συνεδριάσεις λοιπόν είναι αφιερωμένες στην κατανόηση πρώτα ε, του, τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές και από εκεί και πέρα έχουν περιοριστεί σε γενικές αρχές. Θέλουμε τη χώρα ε, προορισμού, ε, θέλουμε την ε, προμήθεια, την αρχή CTP, όχι έτσι. Σε γενικές αρχές κινείται ακόμα η συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο στο Συμβούλιο. Προθυμία υπάρχει να, να συνεχιστούν οι συζητήσεις, αλλά τώρα για το χρονοδιάγραμμα επειδή είναι τεράστιο το εύρος, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να σας δώσω μια ιδέα. Ένα χρονικό ορίζοντα για το πότε θα καταλήξει αυτό στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you very much for that uh, from the... Ευχαριστώ για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. From the e to... Από το ΕΛΚ δεν υπάρχει κανείς για να απαντήσει για να κλείσει τη συζήτηση θα πω αυτό που είπε ο εισηγητής, ότι περισσότερες τροπολογίες ε, δεν είναι επίμαχε και θα ψηφίσουμε στι 22 Ιανουαρίου όπω πρότεινε ο κύριος Βάντεν Κέντελάρε χωρί να προγραμματιστούν ε, ιδιαίτερε ε, καθόλου συνεδριάσεις ε, σκιωδών για τις συμβαστικές. Δείτε το διμερός παρακαλώ με τον εισηγητή αυτό. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα. Να ψηφίσουμε εδώ στις 22 πρώτου και στην Ολομέλεια το Φλεβάρι στο Στρασβούργο. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για τις εκθέσεις αυτές που είχαμε πριν την ψηφοφορία. Τη ψηφοφορία την οποία ε, μεταθέσαμε από τις 9.30 στις 10.30 και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 10.30. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Dear colleagues, welcome. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Πού είναι η Ντανούτα που είδα μαζί μου στη διάσκεψη των Προέδρων. Uh, we can start our vote. Αρχίζει η ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε πρώτα δοκιμαστικά. Αρχίζει η δοκιμαστική ψηφοφορία. One ECR, you try to change the place, maybe. Αλλάξτε θέση παρακαλώ, αν δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Great. Don't worry, no problem. We all did this mistake. Many... Ε, κάνουμε λάθη όλοι, βάζουμε τις κάρτες και ανάποδα καμιά φορά. Λοιπόν, Σταματάει η δοκιμαστική ψηφοφορία και ψηφίζουμε κανονικά για το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου για την αναρμόνιση του καθαρίστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς. Αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. Κανονισμός ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Close. Πέρας. 37 υπέρ. Κανείς κατά και δύο αποχές. Τώρα, θα ψηφίσουμε ε, ε, το αποτέλεσμα που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις για τις διασυνοριακές ε, πληρωμές και συναλλαγές. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Η συγκίτρια είναι κυρία Εύα Μάιντελ. Πέρας. 39 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα θα περάσουμε στη μεγάλη ψηφοφορία για τις εποπτικές αρχές. Πώς θα το πω, αρχίσουμε τη μεγάλη πρώτη ψηφοφορία, τη μεγάλη έκθεση. ΑΙΟΠΑ, ΕΣΜΑ και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Συμβιβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G, συμβαστική πάντα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική GA υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική HA υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική HB υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική IA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική QA Υπερκατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική R Υπερκατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική S Υπερκατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 255 Υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 232 Υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική SA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική δεκτή. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική γιού υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AE υψηλών ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AO, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AP, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AQ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AR, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική ARA, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AS, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική BA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική BD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BE, BF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BH Α, δεν ψηφίσαμε την BE. BE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα BH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BF την ψηφίσαμε. Ναι. Ωραία. Όλα τα κάναμε. BH. BI τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BJ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BK. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BL. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BM. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BTA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BWA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BWB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BWC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BXA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα που είμαστε, CAA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 288, όχι. Έχω παλιά έκδοση του κατάλογου ψηφοφορία. Συμβαστική CC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. C, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 37 ψηφί υπέρ 2 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια τους, στους συνεισηγητές. Θα ψηφίσουμε τώρα την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. 40 υπέρ 2 κατά, χωρίς εποχές. Συγχαρητήρια και πάλι στους συνεισηγητέ. Και περνάμε... Στο θέμα των αγροπιστωτικών μέσων και την ανάληψη και άσκηση μύφιντ ε, ε, θεμαφορικά σε συμβαστική α, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ, μία ψήφος κατά δύο αποχές. Ψηφίζουμε την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 38 υπέρ 2 κατά 2 αποχές. Συγχαρητήρια και πάλι στους δύο συνεισηγητές. Και ψηφίζουμε το σημείο 9 μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος. Συμβαστική τροπολογία Β. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το πρώτο κομμάτι των τροπολογιών, την πρώτη ομάδα τροπολογιών, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά, 20 υπέρ. Οπότε οι υπόλοιπες ομάδες τροπολογιών καταπίπτουν. 85. Ψηφίζουμε την 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική D. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ι, e, ε υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική L εγκρίνεται. Συμβαστική M μη υπέρ εγκρίνεται, συμβαστική νη υπέρ εγκρίνεται, συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική π υπέρ εγκρίνεται, συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική R υπέρ αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική W υπέρ κατά εγκρίνεται, Συμβαστική Χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΓ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΔ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ονομαστική κλίση όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ 2 κατά και μία αποχή. Ψηφίζουμε την απόφαση για την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ 3 Τρεις ψηφίκατα και καθόλου αποχές. Οπότε έχουμε την ενισχυμένη πλειοψηφία για όλα τα θέματα. Συγχαρητήρια στους συνεισηγητές για αυτή την ε, πολύ αίσια διεκπαιρέωση των σημαντικών αυτών θεμάτων. Ο συνεισηγητής ο κύριος Ατμαρκάρα ζήτησε το λόγο και τον έχει. Πρόεδρε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι και για όλες τις εκθέσεις αυτές είχαμε 1440 τροπολογίες. Πάρα πολύ λεπτό θέμα και ευαίσθητο, ε, γιατί έχουμε διάφορες ισορροπίες και διαφορές. Θέλω να ευχαριστήσω τη συγκήτρια, τον Μπορχαρτ Μπάλτς που έκανε το πρώτο τμήμα και τους κοιόδης συγκητές, κυρίως των Πρασίνων, ECR ε, και ALDE. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά που καταφέραμε σε ένα τέτοιο θέμα να ε, βρούμε τόσους πολλούς συμβιβασμούς όπου μπορεί ο καθένας να συμφωνήσει χωρίς να έχει χαθεί η ουσία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και για το αποτέλεσμα. Είναι μια καλή αφετηρία για τις σίγουρα σκληρά διαπραγματεύσεις που επίκυνται με το Συμβούλιο, ε, του οποίου η αντίληψη απέχει αρκετά από τη δική μας. Αλλά ελπίζω να είμαστε εξίσου συμπαγείς και ενωμένοι και να ε, ακολουθούμε στις διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου ε, τους κοινοβουλευτικούς μας στόχους και επιδιώξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να προσυπογράψω το λεγόμενο του κυρίου Κάρας. Δεύτερη φορά κατά το μακρύ κοινοβουλευτικό μας βίο που είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε παρόλο που έχουμε ε, συμπληρωματικέ θα και προσωπικότητε και στυλ. Αυτή η συμπληρωματικότητα λοιπόν των δύο συνεισηγητών νομίζω ότι είναι η συνταγή της επιτυχίας. Γιατί ενωμένη στη διαφορετικότητα καταλήγουμε σε αίσιο πέρας. Ε, δεν ήμουν ανέκαθεν υπέρ του μεγάλου συνασπισμού των δύο μεγάλων κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μερικές φορές όταν Μα ευνοεί, ευνοεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενισχύει τη διαπραγματευτική του δύναμη απέναντι στο Συμβούλιο, γιατί όχι. Νομίζω έτσι θα προσπίσουμε το κοινοτικό ευρωπαϊκό ενωσιακό συμφέρον, μάλιστα μια στιγμή που έχει τρωθεί αρκετά δυστυχώς. Και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όπω και ο Οτμαρ του πάντε και όσου κατέθεσαν τροπολογίε. και νομίζω δεδομένη στις προεργασίες που έχει γίνει ε, και με τις διάφορες συνεισφορές ε, και προσθήκες καταφέραμε να τα λάβουμε υπόψη σχεδόν όλα στην έκθεση με μικρές εξαιρέσεις ε, και για κάποια σημεία που είχαμε κάθετες διαφορές και διαφωνίες αλλά ευτυχώς ήταν ελάχιστα αυτά τα σημεία. Πάντως πρετάνευσε το ίδιο πνεύμα της συνεργασίας. Δεν πρέπει να είστε τόσο καχύποπτοι όταν καταλήγουμε σε μια συμφωνία. Θα ήθελα επίσης να επεκτείνω τις ευχαριστίες μου στους δύο συνεργάτες μας, το βοηθό του ΕΟΤ Μαρκάρας και το δικό μου, γιατί πραγματικά ήταν πολύ αξιόλογο το έργο τους, με τη βοήθεια της γραμματείας της ΕΚΟΝ και τους υπαλλήλου των πολιτικών μας ομάδων. Επίσης, να πω και δύο σχόλια για το περιεχόμενο. Το πρώτο είναι ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι συνεκτική. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να μεφόμαστε τις ε, εποπτικές αρχές ε, γιατί δεν ασκούν τα καθήκοντά τους και να αντιλαμβανόμαστε ότι η διακυβέρνηση των εποπτικών αρχών είναι που δεν τους επιτρέπει ε, το παρόντος να ασκήσουν αυτές, την αποστολή και τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τα, την αποστολή και την, το ρόλο των εποπτικών. Και επίσης προσθέθηκε στο πακέτο η καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και νομίζω ήταν ξεκάθαρη η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στην καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, θα πρέπει να ενισχύουμε τη διακυβέρνηση των εποπτικών αρχών. Η ΔΕΜΗ ουσιαστικά ε, καλοπίζουμε απλώς μια κατάσταση χωρίς να την αλλάζουμε ριζικά. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ανάγκη για πραγματικές αλλαγές. Και πραγματικά επειδή είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος και δεν θα είναι εύκολη θέση του Συμβουλίου, έχουμε μεγάλη πρόκληση. Πάντως ξορκίζουμε την ε, Ρουμανική Προεδρία και τη θέλουμε παρακαλούμε να αναλάβει τις ευθύνες ώστε να καταφέρουμε σε αυτό χρόνο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ θερμά τους δύο συνεισηγητές. Πάντως υπολόγισα το έκβαση της ψηφοφορίας. Ε, η πλειοψηφία ήταν από 93 με 95% η πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκαν οι εκθέσεις. Δεν είναι απλά ευρύς Συνασπισμό ή μεγάλο ε, συνασπισμό ήταν σχεδόν ομόφωνη η μεγαλο συνασπισμο ηταν σχεδον Όλες οι πολιτικές ομάδες συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική επιτυχία. Και φυσικά, χάρη στου συγητές μα προλιάθηκε το έδαφος ε, για να καταλήξουμε σε τόσο ευρία συνένεση, ευρεία συμφωνία, σε τόσο ευαίσθητα μάλιστα θέματα. Αλλά και οι σκιώδεις συγκεκριτές και οι πολιτικές ομάδες συνέβαλαν τα μάλα και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό για την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί μπορούμε πραγματικά να ξεκινήσουμε τις διοργανικέ διαπραγματεύσεις με πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση και με ένα επιπλέον σημείο την καταπολέμηση της νομοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Και τώρα πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, γιατί είναι ακόμα ώρα για να κάνουμε ε, δουλειά. Ξεκινάμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου στις 3 το απόγευμα, λύεται η συνεδρίαση.